Right, Κυρίες και κύριοι, καλώς. Καλώς ορίσατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Παρακαλώ και τα μέλη της γραμματείας και το προσωπικό να σταματήσουν τα κουτσομπολιά και τα ε, πηγαδάκια. Σαν δάσκαλος αισθάνομαι. Έγκριση μερίσια διάταξη έχει μια μικρή αλλαγή στο σημείο 16. Ενταλλαγή απόψε με τον κύριο Πιέρ Κράινμπουλ Έχουν κληθεί τα μέλη της Επιτροπής ΔΕΒΕ να συμμετάσχουν, αλλά δεν θα είναι κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΔΕΒΕ. Αυτά είναι επί του πιεστηρίου τελευταία νέα. Εγκρίνουμε ε, την ημέρησια διάταξη. δεύτερη ανακοινώσει του Προέδρου. Δεν έχουμε τη στιγμή της σύνταξη του κειμένου αυτού ανακοινώσει να κάνουμε. Στο σημείο 10 θέλω να πω κάτι όμως. Θα γίνει και κλεισμένο το θυρών για τη λαϊκή δημοκρατία της Βόρειας Κορέας. Ελπίζω να συμφωνείτε. Μάλιστα, σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών ε, της περασμένης συνεδρίασης. Δύο συνεδριάσεις, 10-11 Ιουλίου και 30 και 31 Αυγούστου. Δεν ξέρω αν έχετε σχόλια. Αλλιώς θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά ε, μέχρι το τέλος συνεδρίασης. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε μια κοινή συζήτηση των σημείων 4 και 5. Το 4 είναι παρουσίαση της μελέτης ε, με θέμα την κατάσταση της εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεση και ελευθέρων συναλλαγών με την Ουκρανία, Γεωργία και Μολδαβία και με έμφαση στην Ουκρανία και στη συστημική ανάλυση των κυρίων τομέων και τη μελέτη με θέμα τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Μελέτε που αμφότερε εκπονήθηκαν κατόπιν ανάθεση από την ΑΦΕΤ. Και το σημείο 5, σύσταση προ το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΑΕΔ σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση εν τη Συνόδου Κορυφή του Νοεμβρίου 2017. Σήμερα λοιπόν θα αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας με την παρουσίαση των δύο μελετών, σημείο 4, πριν περάσουμε στο σημείο 5, έκθεση κυρίας Ανδρή Κέινε και Φλέκενστάιν. Σας ανέφερα κάποιες μελέτες που θα μας δώσουν και την απαραίτητη πραγματογνωμοσύνη ε, για τις εκθέσεις που κάνουμε το 18, καθώς επίσης και αποστολές εκεί. Περιμένουμε να μας ενημερώσουν οι εμπειρογνώμονες εκ των έσω ε, για τη σχέση μας με τις χώρες αυτές και να μας προτείνουν ε, κάποιες συστάσεις πολιτικές ε, και να μας δώσουν βοήθεια για τις κοινοβουλευτικές εκθέσεις. Γι' αυτό έχω καλέσει τρεις εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους για να μας παρουσιάσουν τις μελέτες. Εδώ αριστερά μου κάθεται ο κύριος Μπάρας Γιάραμπικ, ε, εξωτερικό συνεργάτη ε, στο Carnegie Endowment για τη διεθνή ειρήνη και εστιάζει κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ουκρανία και τον αντίκτυπο της σύραξη στην περιοχή και ε, Πέκινα. Εργάστηκε στο Freedom House και είναι η πρώτη μελέτη που θα μας παρουσιάσει εκείνος για τη συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία, Μολδαβία και Γεωργία. Στη δίπλα του κάθεται η κυρία Λέιλα Αλίεβα που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και έχει ιδρύσει το Κέντρο Διεθνών και Εθνικών Μελετών, ένα think tank που εδρεύει στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Προηγουμένως εργαζόταν ε, στο ε, Defense College του ΝΑΤΟ, στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, ε, στην υπηρεσία του ΟΗΕ για ε, την ανάπτυξη και αλλού και θα μιλήσει για το Αζερβαϊτζάν. Και δίπλα κάθηκε ο δόκτωρ Χραντ Κωνστανιάν ε, που είναι ερευνητής στο ΣΕΦ στις Βρυξέλλες, πολύ γνωστός ε, για τις μελέτες για θέματα γειτονίας και σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Επίσης διδάσκει στο Κολέγιο Λεγόπ, στο Κολέγιο Βερσάλιους και θα μιλήσει προφανώς για την Αρμενία. Καλωσόριζω και τους τρεις ομιλητές και τους δίνω το λόγο. Να αρχίσουμε από τον κύριο Γιάραμπεκ. Παρακαλώ. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μιλήσω σήμερα για την εφαρμογή της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης και Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία. Είναι τεράστια η μελέτη ε, και θα προσπαθήσω να μιλήσω κατευθείαν για τα κύρια συμπεράσματα και τις κύριες συστάσεις στα 10 λεπτά και ελπίζω να ε, υποβάλλετε συγκεκριμένες ερωτήσεις εσείς από πλευρά σας. Να ξεκινήσω με το μακροεπίπεδο, την υπογραφή και την την κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία ήταν μια εντυπωσιακή απόδειξη της ε, ήρεμης δύναμης, της απαλής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι γνωρίζουμε ότι μετά τη διεύρυνση την τελευταία υπήρξαν ε, ε, προβληματισμοί σε σχέση με το κατά πόσο θα επηρεαζόταν αυτή η απαλή δύναμη soft power της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ αυτή η ε, Συμφωνία Σύνδεση αποδεικνύει πως όχι. Ε, κινητοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και καλεί τις ε, ευρωπαϊκές χώρες και αυτό παρότι επηρεάζονται από την Ρωσία. Αυτό συνέβη Παρότι η συμφωνία αυτή σύνδεσης δεν προέβλεπε οικονομική βοήθεια του ύψους που δόθηκε στις βαλτικές χώρες, ας πούμε. Ιδιαίτερα για την Ουκρανία η συμφωνία και η κύρωση αυτής ε, είχε μεγάλο αντίκτυπο και επιρροή στις πολιτικές αυτής της χώρας, ειδικά για την Ουκρανία μετά τη ρωσική επίθεση και την προσάρτηση της Κρυμαίας. Δεν υπάρχει πλέον ε, επιλογή ε, πολιτικής, φιλορωσικής πολιτικής, δεν υπάρχει δυνατότητα εξορόπησης και γι' αυτό η επιρροή της δύση έχει αυξηθεί καθώς η Ουκρανία και το Κίεβο δεν έχουν πουθενά να στραφούν αλλού. Και γι' αυτό αυτή η συμφωνία και η εφαρμογή της είναι προτεραιότητα Ιδιαίτερα αν το δούμε αυτό ακόμα και με μεγεθυντικό φακό θα δούμε πως η εφαρμογή θα γίνει παρά όλες τις επικρίσεις. Υπάρχει επίσης μεγάλη όθηση για ολοκλήρωση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στην Ουκρανία και τη Γεωργία και όσον αφορά την κοινή γνώμη η Μολδαβία είναι η μόνη πιο περίπλοκη κατάσταση όπου η ρωσική επιρροή της εξωτερικής πολιτικής δηλαδή της Ρωσίας εξακολουθεί να επηρεάζει την κοινή γνώμη αλλά αυτό ε, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διάβρωση και στην διαφθορά και την κακή διακυβέρνηση της ε, ε, κυβέρνησης και δεν σημαίνει απαραίτητος υποστήριξη για την ίδια τη Ρωσία. Η Μολδαβία είναι επίσης μια καλή ε, περιπτωσιολογική μελέτη, αν και Νωρίς ε, θεωρήθηκε ως επιτυχής ιστορία της ανατολικής εταιρικής σχέσης, όμως είναι μια περίπτωση που θυμίζει ότι αυτές οι συνδέσεις με την Ένωση τελικά μετρώνται με την κοινωνική και οικονομική πρόοδο κάθε χώρας και όχι απαραίτητο με το πόσες νομοθεσίες θα περάσουν, πόσοι νόμοι θα περάσουν ώστε να ε, σηματοδοτήσουν την άφηξη των ευρωπαϊκών στάνταρ. Ιδιαίτερα όσοι εργάζεται, ε, ε, ε, μάλλον υπάρχουν δύο στοιχεία, κυρίως ο, η φτώχεια και ο πατερναλισμός που θέτουν τροχοπέδι στην ευρωπαϊκή πορεία, ιδιαίτερα στις περιοχές της Υπέθρου. Η ευρωπαϊκή βοήθεια κυρίως εστιάζει στις περιοχές της Υπέθρου με πιο διαδεδομένο τρόπο και εστιάζει επίσης στην αποπολιτικοποίηση, την αποκέντρωση και την ενίσχυση των κρατικών δυνατοτήτων μέσω της δημιουργίας των σωστών θεσμών. Η διαφορά με τις, με τις περιοχές της Υπέθρου, ιδιαίτερα όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την οικονομική πρόοδο, είναι πολύ διαφορετική. Τώρα, για την συμφωνία και την εφαρμογή της είναι πολύ νωρίς για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπό της, αλλά οι ειδικοί που μελετούν τις χώρες δείχνουν ότι οι εξαγωγές έχουν ανέλθει από το 25% στο 37% από το 2012 μέχρι το 2016, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινεί γιατί αυτό αυξήθηκε εν μέρη λόγω της ρήξης των εμπορικών σχέσεων με τη Ρωσία. Η Ευρώπη έχει ε, ε, ε, επιβεβαιώσει τη θέση της ως εξαγωγή παραγωγικός ε, εταίρος και φτάνει στο 36% ε, στο σύνολο της χώρας. Η Συμφωνία Σύνθεσης της Γεωργίας δεν έχει τόσο ε, προωθήσει τις εξαγωγές προς την Ένωση, αλλά μαζί με τη βοήθεια της Ένωσης έχει κινητοποιήσει τη γεωργική παραγωγή, που είναι ο πιο σημαντικός τομέας για την οικονομία της χώρας. Σε κάθε χώρα δεν, έχουμε, δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση για την Συμφωνία Σύνδεση και Ελευθέρων Συναλλαγών και δεν υπάρχει αρκετή στήριξη από τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Τώρα, η ευρωπαϊκή βοήθεια ήταν πολύ σημαντική ε, βλέπουμε την ε, βοήθεια, ήταν πολύ αποτελεσματική και βλέπουμε την, ε, την οικονομική σταθερότητα σε όλες αυτές τις χώρες, ιδιαίτερα όσον αφορά την Ουκρανία σε μια πολύ σημαντική χρονική περίοδο. Ταυτόχρονα υπάρχει διαφορά και υπάρχει κάτι που νομίζω πως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να, να το λάβουν πιο σοβαρά υπόψη, είναι η διαφορά ε, με το κόστος συμμόρφωσης που είχε αρχικά υπολογιστεί. Και το επενδυτικό κόστος που συνδέεται με τη συμφωνία σύνδεσης και ελευθέρων συναλλαγών δεν παραμελήθηκε. Οπότε υπήρχαν διαφορετικές προσδοκίες όσον αφορά το κόστος και τα ωφέλη όσον αφορά τη βοήθεια της Ένωσης προς αυτές τις τρεις χώρες. Και διανέφερα ότι ο πραγματικός αντίκτυπος αυτών των συμφωνιών σύνδεσης θα μετρηθεί με την κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Επίσης, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει κάποια αντιστάθμιση για το άνοιγμα του εμπορίου, αυτό το είδος της αντιστάθμισης δόθηκε στα κράτη-μέλη υπό τη μορφή διαρθρωτικών ταμείων και ταμείων συνοχής, που δεν είναι ανοιχτά για αυτές τις χώρες. Τελευταία παρατήρηση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρρωγή είναι βέβαια ότι η μικροοικονομική βοήθεια αρχίζει και μέσω της ε, σταθεροποίησης της μικροοικονομικής, η οποία συνέβη, η λιτότητα συμβαίνει τώρα αυτή την περίοδο, αλλά οι ιδιωτικοποιήσεις δεν συμβαίνουν. Και οι ιδιωτικοποιήσεις δεν συμβαίνουν διότι ε, είναι πολιτικοποιημένα, οι πολιτικοποιημένοι θεσμοί, επικρατεί διαφθορά και στο δικαστικό σύστημα και αυτό δεν μπορούμε πολύ γρήγορα να το αντιμετωπίσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε τη βοήθεια και από αυτή την άποψη. Τώρα, σε σχέση με την Συμφωνία σύνδεση, υπήρξε τεχνική και νομοθετική πρόοδος και στις τρεις χώρες, ιδιαίτερα όμως στη Γεωργία. Οι βασικέ προκλήσει είναι το κράτο δικαίου και οι δικαστικέ μεταρρυθμίσει, καθώ και η έλλειψη πολιτική βούληση για την αποπολιτικοποίηση των θεσμών. Στι τρει αυτέ χώρε υπάρχουν ε, τρει θεσμοί. Υπάρχουν ε, ε, θεσμοί, όπω είπαμε, η εισαγγελία αλλά και τα δικαστήρια που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από του πολιτικού. Και αυτό δεν έχει αλλάξει, αν και τελευταία στην Ουκρανία φαίνεται να γίνεται μια εκβάθρον ε, δικαστική μεταρρύθμιση. Νομίζω πως θα πάρει χρόνο, αλλά είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση αξίζει να τονίσει και να εστιάσει σε, αυτά, σε αυτούς τους θεσμούς από εδώ και στο εξή. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ένα-δυο άλλους ε, παράγοντες, για παράδειγμα το πολύ ψηλό, εξαιρετικό ακραία πολιτική πόλωση δεν υπάρχει διάλογος ανάμεσα στην αντιπολίτευση και την κυβέρνηση των χωρών αυτών. Ε, ε, σε αυτό θα έπρεπε να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες φορές η ευρωπαϊκή προσέγγιση συμβάλλει σε αυτήν την πολιτικοποίηση και την αντίληψη περί ε, αντιπαράθεσης πολιτικής, ιδιαίτερα στη Μολδαβία. Ε, αυτό ούτε ο φιλορώσος πρόεδρος Ντόντον θα ήθελε να τελειώσει αυτή την συμφωνία σύνδεση. Δεν νομίζω πως έχει κανένα σχέδιο, ούτε και τις πολιτικές δυνατότητες να κάνει κάτι τέτοιο. Και εδώ θα κλείσω. Η, τα επιτεύγματα της Ένωσης είναι σημαντικά και επιτυχή, αλλά εύθραυστα. Ε, οι θεσμοί που εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο ε, στις χώρες αυτές είναι διεφθαρμένοι, πολιτικοποιημένοι και χρησιμοποιούν το ρόλο της Ρωσίας στις περιφέρειες αυτές ως ε, μοχλό κινητοποίηση, ε, ε, Επικρίσεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η έλλειψη συνοχής όσον αφορά την δικού τη όρους, την αιρεσιμότητα και αυτό παίζει ρόλο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής βοήθεια προ αυτές τις χώρες. Ε, στην Ουκρανία και στη Μολδαβία εξακολουθούν δεν να δρούν οι Ρώσοι ολιγάρχες και αυτό υπονομεύει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην θεωρηθούμε ότι στηρίζουμε κάποιες κυβερνήσεις μόνο και μόνο επειδή οι ίδιες αυτό αποκαλούνται φιλοευρωπαϊκές. Ακόμα και η Γεωργία επηρεάζεται από του δικούς της ολιγάρχες και υποφέρει από την ε, πολιτικοποίηση έχουν υπάρξει προσπάθειες για μεταρρύθμιση, μια ειρηνική μετάβαση το 2012, η ομαλοποίηση του εμπορίου ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ρωσία και αν ψάχνουμε να βρούμε κάτι δηλαδή που έχει πάει καλά, περισσότερο είναι η γεωργία. Η Συμφωνία σύνδεση και η Βοήθεια η Ευρωπαϊκή φαίνεται να παίξαν σημαντικό ρόλο για τι μεταρρυθμίσει σε αυτέ τι χώρε Ήδη για την Ουκρανία η εξισορρόπηση δεν χρειάζεται πια να γίνεται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Πρέπει να συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει μια ευκαιρία όχι να αλλάξει αυτέ τι χώρε προ το καλύτερο, αλλά έχει και μια ευθύνη. Φέρει ευθύνη ιδιαίτερα όσον αφορά την ευρωπαϊκή βοήθεια και αρρωγή, γιατί ιδιαίτερα για την Ουκρανία δεν είναι άμεση βοήθεια, είναι δάνεια. Ε, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η, εκ νέου και άλλοι τομείς. Χρήματα για τον εξυγχρονισμό αυτών των βιομηχανιών δεν υπάρχουν. Επίση, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τοπικέ πολιτικές εξελίξεις θα παίξουν ε, τελικά πολύ σημαντικό ρόλο, παρα, μάλλον περισσότερο σημαντικό ρόλο από ότι η Ρωσία. Δύο καυγάς περί γεωπολιτικής έχει περιοριστεί και η, γεωργική, η, μάλλον η γεωργιανή εμπειρία δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει πολιτική εδραίωση. Τώρα, όσον αφορά την αποπολιτικοποίηση των θεσμών, μπορεί να έχουμε εκεί κίνδυνο αυταρχισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την εδραίωση των θεσμών αλλά ταυτόχρονα να επιμείνει για δημοκρατικές προδιαγραφές και να ενισχύσει τους θεσμούς. Οι θεσμοί υποφέρουν σε αυτές τις χώρες, οι αυτοί πρέπει να ενδυναμωθούν και όχι τόσο οι ίδιοι οι πολιτικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Γιάραμπικ για την εισήγησή σας. Η δόκτωρ Αλίεβα, δεύτερη για το Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το Αζερβαϊτζάν είναι μια από τις σημαντικότερες χώρες για την Ένωση από την περιοχή. Όχι μόνο λόγω μεγέθους, επειδή είναι κοντά σε τρεις μεγάλες περιφερειακές δυνάμεις, Ρωσία, Τουρκία κλπ, αλλά επειδή διαθέτει και ενεργειακούς πόρους και πιο πρόσφατα υπόγραψε κάποιες συμφωνίες για κάποιους διαδρόμους ιδιαίτερα που αφορούν την προμήθεια φυσικού αερίου και είχαμε πρόσφατα και μια νέα συμφωνία που αφορά το πετρέλαιο και την παροχή πετρελαίου μέχρι το 2050. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα καθορίζουν την επιτυχή σχέση μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Ένωσης σε αυτούς τους τομείς, δηλαδή ασφάλεια ενεργειακή, ασφάλεια τροφοδοσίας και εμπορίου και επενδύσεων σε κάποιες περιοχές. όλα αυτά το Αζερβαϊτζάν και οι σχέσεις του με την Ένωση όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και οι λόγοι είναι εξή. Καταρχάς, είχαμε μία παράλληλη απομάκρυνση του Αζερβαϊτζάν από την Ένωση, παρόλο που το 2006 είχαμε μία ρήτρα για τις σχέσεις με την Ένωση Στι γειτονικέ δημοκρατίε όσον αφορά το σχέδιο δράσης που είχε τότε το Αζερβαϊτζάν. Το 2013 λοιπόν ήδη είχαμε επίσημε δηλώσει ότι το Αζερβαϊτζάν δεν ενδιαφέρεται για την ολοκλήρωση αλλά περισσότερο για μια συνεργασία αμοιβαία και ισότιμη. Το λέω αυτό επειδή ίσως το Αζερβαϊτζάν τότε δεν είδε να υπάρχει αντίστοιχη βούληση από την Ένωση και το 90 είχαν πολλά δραματικά συμβάντα στο Αζερβαϊτζάν. Και από τότε προωθούσε το Αζερβαϊτζάν αυτόνομες, ανεξάρτητες πολιτικές συνεργειακές από την Ρωσία. Πολιτικές υψηλού κινδύνου, υψοκίνδυνε. Πάντως αναζήτησε από την Ένωση μια αμοιβαία απάντηση στα δικά του προβλήματα ε ενέργειας και ασφάλειας κυρίως του Αζερβαϊτζάν, ιδιαίτερα όσον αφορά τον Αγκόνο Καραμπάχ. είχαν την εντύπωση στο Αζερβαϊτζάν ότι η Ένωση δεν προσπίζεται εξίσου και με τον ίδιο τρόπο τις αρχές προάσπιση των συμφερόντων, συνόρων όπως σε άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν απομακρύθηκε το Αζερβαϊτζάν. Ταυτόχρονα αυτό συνεδευόταν από την αντίληψη ότι αποτελεί τον άνεμο κρίκο η Ένωση. Και αυτό επηρέασε τις συμφωνίες όπλων του Αζερβαϊτζάν, ιδιαίτερα μετά από τον πόλεμο με τη Γεωργία, όσον αφορά την Ρωσία, συμφωνίες όπλων με τη Ρωσία. Υπήρχε λοιπόν μία απόκληση από την ανεξάρτητη πολιτική σε σχέση με τη Ρωσία προς μια μεγαλύτερη ισόρροπη σχέση δηλαδή σε σχέση με την Ρωσία και την ηγεσία της. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε και τους παράγοντες που αφορούν την οικονομία του πετρελαίου και την πολιτική, την αντίστοιχη, κάτι το οποίο αναφέρεται επαλλημένως στην φιλολογία για αυτά τα θέματα, ώστε να δημιουργηθούν εδώ κίνητρα για την ολοκλήρωση. Εκτός δηλαδή από το να παρέχουν στους ηγέτες πόρους, οι δυνατότητες ταυτόχρονα επιτρέπουν στον ηγέτη να κινηθεί, να ελιχθεί μεταξύ χωρών και να τηρήσει στις αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της περιοχής που επηρεάζουν τις διαφόρες πολιτικές του. Και ένας τρίτος λόγος βέβαια είναι και το πρόβλημα που αφορά τη σχέση Ένωσης Αζερβαϊτζάν και τον τρόπο με τον οποίο οικοδομήθηκε αυτή η σχέση. Επειδή δεν αντιμετώπισε τα δομικά προβλήματα στις μεταρρυθμίσεις, παραδείγματο χάρη η ενισορροπία μεταξύ κράτους και κοινωνίας, όπως λέγαμε προηγουμένως, αυτό αφήνεται στην πολιτική του πετρελαίου. Εδώ δεν είχαμε επενδύσεις όπως θα έπρεπε στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών όπου αναμενόταν περισσότερες ε, επενδύσεις ακόμα και σε σχέση με τις γειτονικές χώρες. Παρ' όλα αυτά, το Φλεβάρι φέτος ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με ένα συνήθιστο τρόπο. Γιατί δεν είναι συνηθισμένο να παρουσιάζεται ένα εταίρο της Ένωσης με δικό του σχέδιο, ε, σχέδιο το οποίο ήταν προς το συμφέρον του Αζερβαϊτζάν και με το οποίο καλεί τέλο πάντων την Ένωση να συνεργαστούν επίση όρει. Αλλά και στην αρχή των διαπραγματεύσεων ήδη φάνηκαν οι διαφορές σε σχέση με την αντίληψη για την χρήση των πολιτικών σε σχέση με την ασφάλεια και για το θέμα του Καραμπάχ αλλά και για το θέμα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Επίσης, είδαμε ότι αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει περισσότερο ρεαλισμό, πηγαίνοντας αυτές και συμμετέχοντας αυτές τις διαπραγματεύσεις, όμως σε αυτές τις σχέσεις υπάρχει πάντοτε ένας κίνδυνος δηλαδή να χρησιμοποιηθούν αυτές οι σχέσεις με το Αζερβαϊτζάν ώστε η κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν να καταδιώξει την κοινωνία των πολιτών που βασίζεται σε δυτικέ ευρωπαϊκέ αρχέ και ιδιαίτερα την ελευθερία και τι διάφορε ελευθερίε που υπάρχουν. Μέχρι τώρα δεν είχαμε σοβαρές, πολύ σοβαρέ διώξει των ακτιβιστών και υποχώρηση των ελευθεριών. Όμως αυτά τα αναφέρουμε λεπτομερώς όπου υπήρχαν περιπτώσεις και είχαμε την απελευθέρωση δύο ατόμων, αλλά έχουμε αρκετού ακτιβιστές, η πλειοψηφία του δηλαδή βρίσκονται ακόμα στη φυλακή. Για θέματα τώρα πολιτικής και ασφάλειας το Αζερμπαϊτζάν είναι πολύ σημαντική χώρα λόγω ακριβώς της δυνατότητα επιρροή άσχηση επιρροή στην πολιτική της, περιφέρεια, της περιφέρειας περιοχής αυτής. Και υπάρχουν ανεπαρκείς επενδύσεις όσον αφορά τη δημοκρατία και εκεί βλέπουμε ακριβώς το αντίστροφο αποτέλεσμα. Δηλαδή έχουμε τις απαγωγές του Αχτάμ Κταρλή στην ε, Γεωργία του δημοσιογράφου. Βλέπουμε λοιπόν την αντίστροφη επιρροή του Αζερβαϊτζάν στις γειτονικέ χώρες όπου ε, είναι πιο δημοκρατικές και πιο επιτυχημένες όσον αφορά τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος εκτροπής σε αυτές τις καταστάσεις και μέχρι τώρα οι έρευνε δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς. Ξέρω ότι η κοινωνία των πολιτών στη Γεωργία προβάλλει έντονα αυτό το ζήτημα και ζητά τη διερεύνηση για το θέμα αυτού του δημοσιογράφου από το Αζερμπαϊτζάν που, έχει, που έχει φυλακιστεί. Για το εμπόριο, τώρα το Αζερμπαϊτζάν έχει επηρεαστεί κατά πολύ βέβαια από την ε, σημαντική μείωση της τιμής του βαρελιού από τα 150 και βάλει 30 περίπου. Και αυτός επίσης είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την προσέγγιση του Αζερβαϊτζάν με την Ένωση. Χρειάζονται επενδύσεις και αντίστοιχα υπάρχει πίεση για μεταρρυθμίσεις. Παρόλα αυτά, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαφάνεια, τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα σε αυτούς του τομείς, γιατί όσον αφορά την διαφθορά, ξέρουμε ότι είχαμε κάποιες επιτυχίες μέσω της θέσπισης ενός συστήματος που μειώνει την διαφθορά στο χαμηλότερο επίπεδο, όμως υπάρχουν μεγάλες μετακινήσεις και ροές κεφαλαίων που δεν ελέγχονται ακόμα από την κοινωνία. Και ξέρουμε ότι είχαν δεχτεί κάποιες ε, κυρώσεις στο Αζερβαϊτζάν ακριβώς σε δύο οργανισμούς λόγω ακριβώς αυτής της κατάστασης. Και αυτό θα πρέπει να το επιδιώξει η Ένωση. Βέβαια, Οι επαφέ τώρα σε κάποιους άλλους τομεί αποδείχθηκαν επιτυχεί, η διευκόλυνση α πούμε θεώρηση και αντιστοιχή συμφωνία. Θα έλεγα ότι τα προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση, τις υποτροφίες κλπ. είναι πάρα πολύ επιτυχή. Και κάπου εδώ θα έπρεπε να τελειώσω. Αλλά για να αναφέρω και κάποιες συστάσεις, να πω ότι υπάρχουν κάποια θέματα που θα ονόμαζα κόκκινες γραμμές. Κόκκινες γραμμές δηλαδή η Ένωση θα έπρεπε να ζητήσει, να απαιτήσει την απελευθέρωση φυλακισμένων, την ύπαρξη περισσότερων ελευθεριών και να καταστήσει σαφές ότι αυτά είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη μιας ισότιμης στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Δηλαδή θα πρέπει σε αυτό το όραμα να συμβάλλουμε ως να συμβάλλει η Ένωση λέγοντας ακριβώς τι προσδοκεί, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μια ισότιμη συμφωνία ή συνεργασία αν δεν έχουμε ε, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να ζητηθεί αμνηστία για όλες τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και για αυτά τα θέματα θα πρέπει να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα η Ένωση με διάφορα benchmarks και θα πρέπει να θεσπίσει και κάποιες επιπτώσεις σε περίπτωση που ακριβώς αυτές οι ρήτρε της συμφωνίας δεν τηρούνται. Δηλαδή, δεν το δικαίωμα στην Ένωση να εφαρμόσει κυρώσεις. Θα έπρεπε λοιπόν να εφαρμοστούν και οι συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και του ΟΣΑ, ο ΑΣΕ, συγγνώμη, σε σχέση με την εξαγωγή εκλογών. Θα πρέπει επίσης να επιταχύνει η Ένωση τον διάλογο για την απελευθέρωση της θεώρησης και επίσης ε, η συμμετοχή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου άλλο ένα κύριο θέμα και τα θέματα που αφορούν επίσης το ITI και το OGP. Τώρα για την τομεακή συνεργασία θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις τωρινές εξελίξεις στι πολιτικέ, ώστε να μην έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Δηλαδή θα πρέπει η Ένωση να θεσπίσει μηχανισμούς που θα συμβάλλουν στην ε, διαφάνεια στα πλαίσια πάντοτε αυτής της συμφωνίας. Ε, βέβαια θα μπορούσα να πω κι άλλα, αλλά νομίζω θα πρέπει να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Δόκτωρα Λίεβα. Ίσως θα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε στη συνέχεια σε Να συνεχίσετε. Ερχόμαστε τώρα στον τρίτο μα ομιλητή, τον δόκτωρα Χραντ Κωνστάνιν για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Πρόσφατα άρχισε να λειτουργεί η ΕΠΑ για την συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενίας και δίνεται μια νέα όθηση στις δύο πλευρές μετά ε, το ναυάγιο της προηγούμενης συμφωνίας. Στόχος είναι να σφυριλατηθούν πιο στενοί δεσμοί και σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνει και την προθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθεί στις και ανάγκες και ε, καταστάσεις που επικρατούν στις χώρες ανατολικής γειτονίας. Όπως κατοχυρώθηκε αυτό στην αθέρωση Πολιτικής Γειτονίας το 2015. Η συμφωνία αυτή, ΣΕΠΑ, είναι και μια σαφής ένδειξη ότι δεν ε, έχει μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα παιχνίδι μηδενικού αποτελέσματος με τη Ρωσία, αλλά θέλει να διευρύνει ε, τις σχέσεις και να συσφίξει τους δεσμούς της με τις χώρες ανατολικής γειτονίας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας και ε, τέλος να καταλήξω κι εγώ σε κάποιες συστάσεις. Είναι απλή σχετικά η συμφωνία σύνδεσης Αν ήταν η παλιά συμφωνία, αφαιρούμε ε, τη δέσμευση της Αρμενίας για την Ευρασιατική ε, Ένωση και καταλήγουμε στη νέα συμφωνία. Ε, για θέματα δικαιοσύνης, ασφάλειας, άμυνας, κλαδικής συνεργασίας και εμπορίου. Να σας περιγράψω λίγο τα κεφάλαια αυτά υπάρχει ένα κεφάλαιο πολύ ισχυρό για το πολιτικό διάλογο, αντίστοιχο με τα κεφάλαια των συμφωνιών σύνδεσης. Είναι ε, η αντιγραφή του ίδιου του κεφαλαίου από τη Συμφωνία Σύνδεσης στη Νέα Συμφωνία ΣΕΠΑ για τις εμελιώδεις ελευθερίες, για τις εκλογές, περιλαμβάνει διατάξεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό καθώς προετοιμάζεται η Αρμενία να έχει μια σημαντική μετάβαση από το Προεδρικό σε ένα προεδρευόμενο πολίτευμα. Υπάρχει ένα και πολύ, ε, πολύ κεφάλαιο για την εξωτερική πολιτική που περιλαμβάνει και τη δυνατότητα συμμετοχής της Αρμενίας ε, σε, σε αποστολές ΕΠΑ ε, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελευθερία και ασφάλεια ε, περιλαμβάνει θέματα όπως είναι η διαφθορά στη δικαιοσύνη ε, και στους θεσμούς. Περίπου ένα προς ένα αντιγραφή του αντίστοιχου κεφαλαίου στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης. Έρχομαι στην τομεακή κλαδική συνεργασία. Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι διαπραγματευτές κατάφεραν να διατηρήσουν το περισσότερο από το κεκτημένο της Συμφωνίας Σύνδεσης. Υπάρχουν πολύ ισχυρά κεφάλαια για την κλιματική αλλαγή, ε, τα κοινωνικά, τις μεταφορές, την απασχόληση, το περιβάλλον και σε αυτά τα κεφάλαια θα δείτε ότι πολλά από τα στοιχεία του κοινοτικού κεκτημένου που είχε ε, δεχτεί και δεσμευτεί να εφαρμόσει η Αρμενία στην προηγούμενη συμφωνία που δεν ευωδόθηκε, διατηρούνται. Υπάρχουν επίση κεφάλαια για την περιφερειακή συνεργασία και την κοινωνία των πολιτών. Ένα κεφάλαιο που είναι κάπως πιο ρηχό έχει να κάνει με την ενέργεια και ιδιαίτερα με το φυσικό αέριο, αλλά και ε, πυρηνικό εργοστάσιο. Ε, το κεφάλαιο για το εμπόριο είναι εκείνο που θίγεται περισσότερο από τη συμμετοχή της Αρμενίας στην Ευρωασιατική Ένωση. Δεν είναι προτιμησιακή η σχέση και το καθεστώς που δίνεται στην Αρμενία. Δηλαδή δεν ε, καταργούνται οι δασμοί εκατέρωθεν. Εξού και είναι ρηχό το κεφάλαιο και, και φτωχό. Ε, από την άλλη όμως ε, υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις για, την, για το καθεστώς γενικευμένων προτιμήσεων συν. Και κάποια κεφάλαια για τα τελωνιακά ζητήματα έχουν να κάνουν με τη ιδιότητα του μέλους της Ευρωσιατικής Ένωσης. Από την άλλη, οι διαπραγματευτές κατάφεραν να καταλήξουν σε ένα καλό κεφάλαιο για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις. Η Αρμενία θα συνεχίσει να είναι μέλος της Ευρωσιατικής Ένωσης, αλλά θα έχει ένα, μια ρυθμιστική αρχή σαν αυτούς που διαθέτουν χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίση, υπάρχουν και άλλα στοιχεία στο εμπόριο, οι υπηρεσίε, που είναι το ουσιαστικότερο τη σημερινή συμφωνία, αλλά και ε, δημόσιε ε, συμβάσεις και ε, θέματα πνευματική ιδιοκτησίας. Από το 2013 η Αρμενία ήταν στην ίδια ομάδα με το Αζερβαϊτζάν και τη Λευκορωσία χωρίς συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Αυτό όμως το αφήγημα παραγνωρίζει την ε, ε σημασία της νέας συμφωνίας και την υποβαθμίζει. Μετά την επιτυχή ε, διαπραγμάτευση θα πρέπει να περάσουμε τώρα σε μια επιτυχή υλοποίηση τη τη Προχωρώ στάση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τονίσει πόσο σημαντικός είναι ο πολιτικός διάλογος. Το Κοινοβούλιο να επικεντρωθεί στις μεταρρυθμίσεις ε, των ε, αρχών επιβολής του νόμου να προχωρήσει το σχέδιο δράσης για την απελευθέρωση ε, θεωρήσεων καθώς η Αρμενία έχει επιτυχώς εφαρμόσει τη Συμφωνία Διευκόλυνσης ε, Θεωρήσεων και τη Συμφωνία Επανεισδοχής, οπότε δεν υπάρχει ουσιαστικό εμπόδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να υλοποιεί το σχέδιο δράσης για την απελευθέρωση θεωρήσεων και να επιζητά αυτήν. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμμετέχουν καλύτερα οι μη ε, κρατικοί φορείς στην εφαρμογή της συμφωνίας και τέλος θα πρέπει να ενισχυθεί η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινωνία των πολιτών και στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και στη μεταρρύθμιση του δημοσίου αλλά και ε, της δικαιοσύνης. Σταματώ εδώ για να έχουμε περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δόκτωρ Κωνστανιάν. Ακούσαμε τους τρεις προσκεκλημένους ομιλητές μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στα μέλη που επιθυμούν να κάνουν ερωτήσεις. Θυμίζω, μάλλον ότι θέλω να σας πω το εξής. Αν θέλετε να αναφερθείτε στο σχέδιο έκθεσης θα πρέπει να περιμένετε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Τώρα ζητούμε το σημείο 4. Ερωτήσεις που έχουν άμεση σχέση ε, με τα όσα ακούσαμε. Έχω εδώ ένα κατάλογο μιλητών. Αρχίζουμε. Πρώτος ο κύριος Σόλτς. Παρακαλώ, Χέλμουτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Um, Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές για την ενημέρωσή τους ε, τόσο εμπεριστατωμένη. Ε, κύριε Γιάραμπικ, μιλήσατε για κάποιες δομές ολιγαρχών που εξακολουθούν να ε, κυβερνούν εκεί παρά τα επιτεύγματα. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό, για ποιους λόγους γίνεται αυτό στη Μολδαβία, στην Ουκρανία, Ιδιαίτερα αναφερθήκατε όμως και στη Γεωργία. Γιατί παραμένουν τέτοιες δομές και έτσι έχει η κατάσταση ότι ε, αυτές οι ολιγαρχικές δομές επηρεάζουν τόσο πολύ, κυριαρχούν στην οικονομία ενδεχομένω και στις πολιτικές εξέλιξεις. Μια ερώτηση προς την κυρία Αλίεβα. Και στον κύριο ε, δεν άκουσα ιδιαίτερα για τον Αγκόρνο Καραμπάχ μια πρόταση. Τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο ρόλο να διαδραματίσει εκεί για να ξεπεραστεί αυτή η σύγκρουση. Είναι μια συνεχιζόμενη σύγκρουση και είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ και τις δύο χώρες με την προσωπία της Επιτροπής ΑΦΕΤ και είδαμε ότι η σύραξη στον Αγκόρνο Καραμπάχ είναι ένα θέμα φλέγων και για τις δύο κοινωνίες και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενέχεται άμεσα αλλά με την συμφωνία σύνδεσης, με τις άλλες πολιτικές επαφές και την οικονομική συνεργασία θα μπορούσαμε ενδεχομένω να συνεισφέρουμε έτσι ώστε να υπάρξει ή να διαμορφωθεί μια τέτοια κατάσταση εσωτερική ώστε να υπάρξει προθυμία να ξεπεραστεί να λυθεί αυτό το θέμα. Ευχαριστώ εξαιρετικές ερωτήσεις. Και εγώ πραγματικά χάρηκα που δεν άκουσα να φέρτε τον Αγκόνο Καραμπάχ, αλλά το ήξερα ότι κάποιο θα το ανέσυρε. Στο μεταξύ έχουμε αρκετού συναδέλφου που ζητούν το λόγο. Θα σας πρότεινα να ακούσουμε πρώτα τις ερωτήσεις και μετά να μοιραστείτε τις απαντήσεις. Ποιος θα απαντήσει σε ποια ερώτηση. Τώρα μεγάλε μεγάλες πολιτικές ομάδες ξύπνησαν. Ο κύριος Στέτινα. E, Σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ναι, βάλτε καλύτερα τα ακουστικά σας παρακαλώ. Το ερώτημά μου ε, το απευθύνω στον κύριο Κωνστανιάν. Με ακούτε παρακαλώ. Τάσκα. Never mind, I will, I will ask in English. Με ακούτε κύριε Κωνστανιάν. Eh, Ωραία, να ξαναρχίσω. Κύριε Κωνσταντιάν, ελπίζω τώρα να με ακούτε. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αναφέρατε την απελευθέρωση των θεωρήσεων για την Αρμενία. Γιατί να μην το συγκρίνουμε με την ε, Γεωργία και τη Μορδαβία που ήταν μεγάλη ε, επιτυχία. Ποιες προθεσμίες ε, σκέφτεστε, δηλαδή πότε πιστεύω ότι μπορεί να γίνει η απελευθέρωση για την Αρμενία. Φλέγκεστάιν. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Μία ερώτηση θέλω μόνο να κάνω σε σχέση με την πρώτη ομιλία για τους ολιγάρχες που αναφέρατε. Σωστά είπατε ότι στη Μολδαβία θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τι συμβαίνει. Ακριβώς γιατί ο πρώτος αυξάνει όλο και περισσότερο την εξουσία του και ο δεύτερος είναι φυλακή. Οπότε, είπατε ότι σε ό,τι αφορά τη γεωργία, αν σας κατάλαβα καλά, το θέμα είναι μάλλον υπηότερο γιατί είναι πολύ περισσότεροι και ολιγάρχες. Για την Ουκρανία Σιγή τι έγινε, το λύσανε εκεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, Κνούτ Φλέκενστάιν. Και τώρα η κυρία Λαλόντα από τους Φιλελευθέρους. Oui, Monsieur Μάλιστα, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήθελα απλώς να να μιλήσω για την έκθεση για το Αζερβαϊτζάν. Έγινε λόγος για την κοινωνία των πολιτών και συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Λίεβα. Όμως, σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών, πιστεύω πως είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να υπογραμμίσουμε, είναι τα γυναικεία δικαιώματα. Έχω για την ευκαιρία να βρεθώ επανειλημμένα στο Αζερβαϊτζάν και πρέπει να πω ότι είναι ε, ασκείται μια πολιτική υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών. Είναι εξαιρετικό το τι συμβαίνει εκεί. Ήμουνα στα σύνορα ανάμεσα στο Αζερβαϊτζάν και το Ιράν και γίνεται μια πολιτική για να καταπολεμηθεί να καταπολεμηθούν οι παιδικοί ε, γάμοι που είναι εξαιρετικοί. Εγώ λοιπόν έχω πολύ περιπλανηθεί στο Αζερβαϊτζάν, σε περιφέρει, κοντά στον Αγκόρνο Καραμπάχα, ε, είδα την πολιτική που ασκείται απέναντι στους εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες και νομίζω πως είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τα ισχυρά σημεία. Εγώ ήμουν εκεί, ε, έκανα αποστολές, εκεί είναι εξαιρετική περίπτωση, είναι 85% μουσουλμάνοι και όλες οι επαρχίες ε, έχουν νούμερο ένα γυναίκα, αν όχι είναι νούμερο δύο η γυναίκα. Ε, είναι σημαντικό να το λέμε και αυτό και εφαρμόζουν ε, το ψήφισμα του ΟΗΕ για τις γυναίκες που πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχουν ε, παντού ε, ενημερωτικά προγράμματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι ασκείται αυτή η πολιτική υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτσης. Uh, οι συμφωνίες αυτές δεν μπορούν να παραβλέπουν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αρχές και ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάρτηση των διακρίσεων κτλ. Και να πω και κάτι για την Μολδαβία γιατί δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε καλά νέα για αυτά τα θέματα, επίσης και για τις προμήθειες ε, του δημοσίου. Έχουμε θέματα που αφορούν τη ελευθερία των ΜΜΕ, τις τράπεζες, ο έλεγχος των ΜΜΕ. Υπάρχουν εκεί που λένε ότι ελέγχονται τα ΜΜΕ, έχουμε αύξηση της καταστολής και αυτό γίνεται με κάποιους έτσι αφιλεγόμενους τρόπους. Αυτή λοιπόν η κατάσταση πώς επηρεάζει την εφαρμογή της ΕΠΑ. Επίσης, όσον αφορά τη χρηματοδότηση της Μολδοβίας από την Ένωση, όταν λέμε ότι λειτουργούν και είναι αποτελεσματικές αυτές οι συμφωνίες δεν θα πρέπει μόνο να επικεντρωνόμαστε στα οικονομικά ζητήματα, αλλά και στα κοινωνικά και στα ζητήματα ελευθεριών. Ευχαριστώ. Χάουταλα και Πίτσουλα. Και μετά θα δοθούν οι απαντήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Ο κύριος Ιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης. Νομίζω ότι δεν αναφέρθηκε σε κάποια πράγματα και τον παραθέτω. Θέλω τώρα να ενισχύσουμε την ατζέντα για το εμπόριο. Υπάρχουν διάφοροι εμπορικοί εταίροι οι οποίοι συνοστίζονται στην πόρτα μας για εμπορικές συμφωνίες και τέλος η Ευρώπη θα πρέπει πάντοτε να πρασπίζει τα στρατηγικά της συμφέροντα. Τέλος της παράθεσης. Αναφέρθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Αφρική, στα Βαλκάνια, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Νέα Ζηλανδία. Αλλά δεν μιλήσε για τις χώρες που συζητάμε σήμερα. Υπό το φως βέβαια των εμπορικών συμφωνιών. Οπότε ρωτάω. Έχετε σχολεία γι' αυτό. Πώς σας φαίνεται. Θεωρείτε ότι η εταιρική μας σχέση με αυτές τις χώρες είναι εκτός πεδίου ένωσης ή εκτός τέλο πάντων πεδίου των σχεδίων της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η κυρία Χάπταλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δυστυχώ και εγώ θα πρέπει να αναφερθώ στο Ναγκόνο Καραμπάχ που είναι τόσο οδυνηρό ζήτημα για όλη την περιοχή και για τις σχέσεις μας με την Ανατολική Εταιρική Σχέση και χώρο όπως το Αζερβαϊτζάν με την Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω πώς η Ένωση Κύριε Κωνσταντιάν, ακούστε με, για εσάς ε, είναι η ερώτηση, για ακούστε με λίγο. Δεν αφήσαμε εκτός αυτή τη συζήτηση, αυτό το θέμα αυτή τη συζήτηση, αλλά να μου πείτε πραγματικά ποια θα ήταν η μόχλευση της Ένωσης για την ειρηνική επίλυση αυτού του ζητήματος. Επειδή ξέρω ότι αυτή τη στιγμή την... ότι έχουμε συμφωνία την ΣΕΠΑ που είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε την Αρμενία. Έχουμε και τη νέα συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν. Οπότε έχει διαθέτει η Ένωση αυτή την απαραίτητη μόχλευση. Είναι απαραίτητο, είναι καλό να αναφέρουμε το ομάδα του Μίνσκ σε αυτό το θέμα. Και να συνεχίσω. Θεωρείτε ότι υπάρχει έλλειψη συνέπειας ή δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εκ μέρους της Ένωσης εδώ μιλάει για έλλειψη κυριαρχία σε περίπτωση Μολδαβίας, ε, Ουκρανίας κτλ. Αλλά δεν μιλάει για Αζερμπάτζαν και Ναγκόνο Καραμπάχ με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, συνάδελφοι, θα έλεγα να δώσουμε στον κάθε εισηγητή πέντε λεπτά για να απαντήσει όσο μπορεί. Απλά και μόνο να αποφασίσουμε τώρα ποιος θα απαντήσει πρώτος. Πρώτα οι κυρίες θα έλεγα, αλλά δεν θα ήθελα να παρενεύω έτσι σε αυτή τη σχέση Αρμενίας Αζερβαϊτζάν. Θέλετε εσείς πρώτα? Ναι. Ναι, θα το κάνουμε να Καρμπάχ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Οι ολιγάρχες αυτές της περιοχής, κυρίως στην Ουκρανία, δεν τους ανέφερα επειδή δεν είναι ότι δεν διαρματίζουν σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα μάλιστα στην Ουκρανία, αλλά γενικά τονίζουμε υπερβολικά τον ρόλο αυτών των ανθρώπων. Και οι ολιγάρχες εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να τους ονομάσουμε οικονομικές πολιτικές ομάδες σε σχέση με το κράτος. Μετά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης είχαμε την, τις ιδιωτικοποιήσεις, τα ξέρουμε όλα αυτά, αλλά ανέκυψαν αυτές οι ομάδες επιρροής. Το θετικό με αυτού είναι ότι όταν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ του όπως στην Ουκρανία ή όπως είχαμε στην ε, Μολδαβία, τότε έχουμε μια ισορροπία, η οποία προέρχεται από αυτούς προερχεται απο αυτου από το κράτο. Τώρα για τις συμφωνίες αυτές η κατάσταση είναι διαφορετική. Η Ένωση ε, ήρθε στην περιοχή το 4 με τις διευρύνσεις. Μιλάμε για 13 χρόνια παρουσίας εδώ. 13 χρόνια. Γι' αυτό μιλάω για μια σημαντική επιτυχία όσον αφορά αυτά τα 13 χρόνια. Κανείς εδώ δεν θα ήξερε που ήταν η Ουκρανία ας πούμε, στον ε, πολιτικό χάρτη ή ούτε καν η Λευκορωσία μάλιστα ούτε κυριοφορουσία. Και αυτό βεβαίω έχει να κάνει με το θέμα των λιγαρχών και θα έλεγα ότι με, την, με τη συμφωνία σύνδεση, οι οποίε ενισχύουν βεβαίω τα κράτη αλλά τα απολυτικοποιούν, Και έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία που θα δείτε στην έκθεσή μας και βλέπουμε ότι οι ολιγάρχες και σιγά σιγά το πρόβλημα που τους συνοδεύει θα εξαφανίζονται, υποχωρούν λόγω ακριβώς των ε, πολιτικών δυναμικών έχουν δεχτεί σημαντικά πλήσματα. Ο Σαχμέτοφ, ο οποίος είναι ο πιο α, ε, από αυτούς. Είχαμε την... Έχουμε τις περιουσίες οι οποίες υποχώρησαν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια λόγω σειράξεων, λόγω κατέθεση τη Ουκρανία κτλ. Και παρόλο που ο πρόεδρο είναι και αυτό ο Λιάρχη, υπάρχει κάποια ισορροπία μεταξύ τέλο πάντων τη ενίσχυση των θεσμών του κράτου, τη ανοικονόμηση του κράτου, του κοινωνικού συμβολέου και των δυτικών συμφερόντων που είναι πάντοτε παρόντα. Νομίζω ότι η Ένωση ακριβώ θα πρέπει να επικεντρωθεί στη σύγκρουση συμφερόντων που αφορά και του ολιγάρχε, αλλά και τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα που εκπροσωπούνται. Αλλά η Ένωση εδώ δεν μπορεί να κάνει κάτι για να το εξαφανίσει. Η Γεωργία είναι κάπως διαφορετική περίπτωση. Γιατί θυμάστε το Κασβίλη και ε, θυμάστε ότι εισήλθε σε αυτές τις πολιτικές κάπως αργά. Έχουν εξελιχθεί τα πράγματα πάρα πολύ πριν 10 χρόνια τον ήξερα, ήταν κάποιο πλούσιο. Κάποια στιγμή περίμενα να θα μπει στην ε, πολιτική γιατί ε, έχτιζε παλάτια τέλο πάντων σε πολύ γνωστά μέρη κτλ. Αλλά όλα αυτά βοηθούσαν και την δημοκρατική μετάβαση της Γεωργίας. Έχουμε πάντως σήμερα τα Γενικό Εισαγγελέα και τη δικαιοσύνη, έχουμε και τις ε, μυστικές υπηρεσίες στην περίπτωση της ε, Ουκρανίας και αλλού που πραγματικά καταδιώκουν αυτούς τους ε, ολιγάρχες και η θέση τους έχει υποχωρήσει. Θα έλεγα λοιπόν ότι όλο αυτό οφείλονται και στις δικαστικές μεταρρυθμίσεις, ε, οφείλονται στο Γενικό Εισαγγελέα και όλα αυτά νομίζω θα έπρεπε να αποτελούν μεγαλύτερο σημείο εστίασης για την Ένωση και όντως είναι ώστε να δοθεί περισσότερη εμπιστοσύνη δηλαδή στις αρχές αυτές, αυτές τις χώρες ώστε να προχωρήσουν. Και το άλλο για το ρόλο των μέσων που δεν υπογράμμισα αλλά επικεντρώνεται η μελέτη στο θέμα των μέσων σημαντικά για την ιδιοκτησία ακαθόδε ζήτημα και στις χώρες μέλη της Ένωσης και δεν νομίζω ότι ας πούμε η κατάσταση στα μέσα της ε, Ουκρανίας που είναι ισορροπημένη όσον αφορά στους ολιγάρχες διαφέρει πολύ από το Ηνωμένο Βασίλειο έτσι για καμία σύγκριση. Οι ολιγάρχες βεβαίως είναι οι ιδιοκτήτες αλλά υπάρχει κάποια σχετική ισορροπία και η άλλη διαφορά είναι και τα κρατικά Ε. Ποιος είναι ο ρόλος των κρατικών ΜΜΕ. Και νομίζω ότι εδώ ακριβώς θα έπρεπε να εστιάσουμε ως μεταρρυθμίσεις και το κάνουμε στην έκθεση. Σχετικά τώρα για το λόγο του κύριου Γιούνκερ δεν μπορώ να σχολιάσω. Δεν ξέρω γιατί έλειπε η ανατολική εταιρική σχέση από το λόγο του. Νομίζω πάντως ότι η Ένωση αυτή τη στιγμή εξετάζει την ανατολική εταιρική σχέση μέσω αυτών που συνέβησαν τα δύο τελευταία χρόνια όπου είχαμε μια κατάσταση πολέμου στον Τόμπας. Και αν το δούμε σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, νομίζω η εικόνα θα είναι διαφορετική. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχει αναφερθεί η ανατολική εταιρική σχέση και θα πρέπει η Ένωση να το εξετάζει περισσότερο. πέρα από 30 χρόνια δεν υπήρχε Ένωση, οπότε έχουμε διανύσει τεράστια απόσταση, εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια, αλλά και η Ευρώπη νομίζω θα πρέπει να εμπλακεί με περισσότερη ευθύνη και παρουσία στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη και κύριε Αλίεβα τώρα. Βασικά δύο θέματα με ρωτήσατε. Το ένα αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Θα πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα δεν είναι παρά μια μικρή αντανάκλαση, μια μικρή ένδειξη του τεραστίου δυναμικού ε, των γυναικών και των δικαιωμάτων τους και τις γυναίκες σε θέση εξουσία. Τι γίνεται με τις γυναίκες στο Αζερβαϊτζάν όταν έχουμε απελευθέρωση, πότε έγινε αυτό. Πολλοί μίλησαν για τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, όταν δημιουργήθηκε το λαϊκό μέτωπο και το πιο δύσκολο έργο το είχαν αναλάβει γυναίκες, ε, τότε που υπήρχε κενό, κενό εξουσίας. Ε, κατάφεραν να χειριστούν τα πιο δύσκολα γαθήκοντα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Η γιαγιά μου ήταν πρώτη πτυχιούχος ε, του πρώτου κοσμικού σχολείου για μουσουλμάνες. Ε, όπου ε, από εκεί ξεκίνησαν ε, διάφορες γυναίκες που έγιναν και εκατομμυριούχοι στις αρχές του 20ου αιώνα και στη συνέχεια συνεισέφεραν πάρα πολύ στην ανάπτυξη της χώρας. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα τι μπορούν να κάνουν οι γυναίκες στην κοινωνία του Αζερβαϊτζάν. Είχαμε μια πολύ ισχυρή παράδοση απελευθέρωση της γυναίκας ε, πριν τη Σοβιετική εποχή, διαστρεβλώθηκε λίγο επί ε, Σοβιετικής ε, εποχής και τώρα δυστυχώς κάπως πιέζεται αυτός ο κοσμικός χαρακτήρας. Για τον Αγκόρνο Καραπάχ δεν κάναμε κάποιες κοινέ συστάσεις. Βεβαίως ο καθένας έχει την άποψή του για το πώς θα μπορούσε να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά θα έλεγα ότι είναι ανεπαρκής η παρουσία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στα πλαίσια ε, των παγκοσμίων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δυτικές χώρες, τα δυτικά κράτη απέναντι σε αυταρχικά κράτη. Είναι σημαντικό, γιατί έχουμε τη Ρωσία που είναι πολύ πλεγμένη σε αυτή τη σύγκρουση. Και όσο παραμένει εκεί ε, α, χωρίς να την αντιμετωπίζει κανείς, τόσο αναπτύσσεται και ο αυταρχισμός στις χώρες μας. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Είναι ένα τρίγωνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως ξέρουμε ότι είναι μια ήπια δύναμη. Αυτή είναι και η, αξία της, και η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχω ξαναπεί και την περασμένη φορά. Ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν διακρίσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων μειονοτήτων. Γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος σε σχέση με αυτά. Όπως είπε η κυρία από τη Φινλανδία, η κυρία Χάουταλα, υπάρχει μια αίσθηση στον φιλανδια Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικά οποιοδήποτε μεσολαβητής ε, προσεγγίζει το θέμα με κριτήρια πολιτιστικά και πολιτισμικά σε αντίθεση με άλλες συγκρούσεις. Κάτι άλλο που θεωρώ πολύ θετικό. Υπάρχει μια τάση που διαπιστώσαμε στην περιοχή. Μόλι ολοκληρώσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για να δούμε πώ αντιδρά ο ενεργός πληθυσμός. Δεν υπάρχει κανένα ε, βασικό μίσος ε, ε, έτσι, πρωταρχικό. Σε αντίθεση με τις μαζικές μελέτες που δείχνουν ότι ο κόσμος έχει πολύ αρνητικά αισθήματα ο ένας προς τον άλλον, λαοί κτλ. Αλλά βαθύτερα αν το ψάξετε θα δείτε ότι αναδύεται μια νέα γενιά που προσπαθεί να ξεφύγει ε, από τις ε, παλιές αντιλήψεις, να περάσει προς τη σύγχρονη εποχή ε, και να βρούμε μια λύση. Γιατί από τη μια έχουμε το διεθνές δίκαιο που είναι στο πλευρό του Αζερβαϊτζάν, είναι τέσσερα τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, από την άλλη έχετε το ε, στατιωτικό status quo, την πολιτική επιρροή της Αρμενίας στην Δύση, δηλαδή έχετε από τη μια την Real πολιτική και από την άλλη την, διεθνή νομιμότητα. Πώς θα καταλήξει ένα συμβιβασμό, γιατί και οι δύο θέσεις ε, έχουν πολύ ισχυρά ερίσματα. Από την άλλη όμως βλέπετε ότι ε, μεγαλώνει μια νέα γενιά ε, που ζει σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο και τον βλέπει σε πολύ διαφορετικό επίπεδο αυτό το θέμα, αυτή τη σύγκρουση. Με διαδικασίες ένταξης όταν τα σύνορα δεν θα είναι κάτι το αδιαπέραστο. Υπάρχουν πολλές λύσεις και άλλα παραδείγματα από άλλες καταστάσεις και μπορεί αυτή η σύγκρουση να ε, αλλάξει και να ανοίξει μια νέα διάσταση. Αυτή είναι η άποψή μου. Um, ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Κωνσταντιάν. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω κάτι που μόλις ανέφερε η Αλέιλα, την, την ε, αποφασιστικότητα και τη στήριξη Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό. Τώρα τα ψηφίσματα, αν τα διαβάσετε βεβαίως, πάντα λένε, καλούν για πάυση πυρός. Και αυτό δεν το εφήρμοσε το Αζερμπαϊτζάν. Θα δείτε δηλαδή ότι υπάρχει μία εφαρμογή και από τις δύο πλευρές. Η κυρία Χάουτλα μόλις έφυγε ή μίλησε για διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Δεν νομίζω πως τίθεται τέτοιο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομιζω οτι υποστηθεται διαφορετική προσέγγιση απέναντι σε διαφορετικές ε, ε, συγκρούσεις. Από τη μια πλευρά βλέπουμε ότι δίνει προτεραιότητα στην ακυρεότητα την εδαφική, ενώ στην άλλη πλευρά την αυτοδιάθεση, αν δούμε πούμε, το κοσφοπέδιο. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση σε αυτές τις συγκρούσεις και όχι μόνο για τις χώρες. Έχουν διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές ε, παράγοντες. Ε, ας πούμε, η Ρωσία συμμετέχει σε πολλές συγκρούσεις, αλλά όχι άμεσα σε αυτήν του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα από αυτά που κάνει, αλλά όχι να δικαταστήσει την, ε, την ομάδα του ΜΙΣΚ. Και με εξέπληξε που θέσατε τόσα πολλά ερωτήματα για τον Αγκόρκο Νότα Καραμπάχ, αλλά όχι για τον Ντομπάς, ούτε για την Κρυμαία. Ε, να πω δύο λόγια για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον των προσπαθειών που γίνονται για βοήθεια ή στήριξη της ομάδας του Μίνσκ. Η η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ας πούμε να καταδικάζει την στρεβλή διτητορία και να καταδικάζει τις ενόπλες συγκρούσεις. Μπορεί επίσης να προωθήσει ένα μέσο ή ένα μηχανισμό ώστε να βρει ακριβώς τι συμβαίνει επί τόπου. Μπορεί να απαιτήσει ο ειδικό εκπρόσωπος της ε, να εφαρμόσει την εντολή του πλήρως. Και βεβαίως μπορεί να ε, ξεκινήσει με, και, να, και να έχει επαφές με ουδέτερο τρόπο με το λαό του Νακόρνου Καραπάχ. Αλλά θα πρέπει να χάνει και το δημοκρατικό της στόχο, γιατί τα δημοκρατικά κόμματα εκεί θα μπορέσουν να βρουν πολύ πιο εύκολα λύση από ότι χώρες οι οποίες είναι αυταρχικές. Απελευθέρωση θεωρήσεων. Πολύ σύντομα είναι πολύ δύσκολο να πούμε πόσο μπορεί να πάρει η απελευθέρωση. Αν δούμε διαφορετικέ χώρε, Μολδαβία, ε, σε αντίθεση με την Ουκρανία, βλέπουμε διαφορετικού χρονικού ορίζοντε. Το πιο σημαντικό όμω είναι να αρχίσει κάτι. Και μετά είναι μια διαδικασία. Εξαρτάται πόσο καλά θα τα πάει κάθε χώρα. Αν η Αρμενία πούμε, προχωρήσει καλά στο αναμαθητικό του επιτυχίο, ε, τότε μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα. Υπάρχουν διάφορα blog, διάφορες εκθέσεις, υπάρχουν ε, τεχνικές μελέτες και παραμένει και η πολιτική απόφαση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ξεκινήσει η απελευθέρωση και τώρα πόσο καιρό θα πάρει θα εξαρτηθεί από τα μέρη. Γιατί έχουμε και θέματα ε, διαφθοράς που είναι πολύ σημαντικά σε αυτή τη φάση. Κυρία Λίεβα, κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστούμε για τις δηλώσεις και για το απαντήσατε, που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Καλείστε αν θέλετε να παραμείνετε, γιατί έχουμε μια επόμενη συζήτηση για αυτές τις χώρες. Και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θα ήθελα να εξετάσουμε για δεύτερη φορά το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Αντρικένη και του κυρίου Φλέγκεστάινα εν ώψη της ε, Συνόδου Κορυφής του Νοεμβρίου του 2017 και σε σχέση με συστάσεις του Συμβουλίου, ε, τη σύσταση μάλλον προς το Συμβούλιο. Η προηγούμενη εξέταση της έκθεσης ήταν στις 14 Ιουλίου στο Στρασβούργο Και τώρα είμαστε στη δεύτερη εξέταση της έκθεσης. Θα δώσω στους δύο εισηγητές το λόγο. Η κυρία Άντρη Κένε, θέλετε να ξεκινήσετε. 5 με 7 λεπτά και μετά ο κύριος Φλέγγεστάιν και μετά μια σύντομη συζήτηση. Αν θέλετε εσείς να ξεκινήσετε, παρακαλώ Κνούτ. Εναλλάξει, την τελευταία φορά άρχισε πρώτα η συνάδελφος, τώρα εγώ και μετά ξανά η κυρία Ανδρικένε. Αυτό είναι και μια ένδειξη πολύ καλής συνεργασίας. Μπορεί να μην συμφωνούμε αυτόματα σε μερικές λεπτομέρειες, πάντως μπορούμε πάντα να βρίσκουμε συμβιβασμούς, είτε επί της ουσίας, είτε γενικότερα. Όταν γνωρίζουμε ότι κάποια θέματα δεν είναι του παρόντος και μπορούμε να τα αφήσουμε για ευθετότερο χρόνο. Δεν χρειάζεται να τονίζουμε τις διαφορές και να τις προβάλλουμε όταν είναι δευτερεύουσες, αλλά τα όσα μας ενώνουν. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ την συνεισηγήτριά μου και τους σκιώδης ηγητές και όλους τους υπολείπους συναδέλφους που με τις τροπολογίες τους βοήθησαν και συνεισέφεραν ε, στην παρούσα έκθεση. Ποιο είναι το βασικό και κεντρική ιδέα της έκθεσης. Δεν θέλω να μπω τώρα σε όλες τις λεπτομέρειες. Σίγουρα τα διαβάσατε όλα σε πολλές λεπτομέρειες. Η κεντρική ιδέα ήταν εξή. Η παράγραφη ε, Χ ε, ψη και ε, ο συμβιβασμός 26. Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία. Οι τρεις αυτές χώρες έχουν κάνει και πολύ ε, λόμπι με τη θετική έννοια, με την καλή έννοια. Ε, για να πάρουν ε, μια προοπτική ε, ένταξης. Και θέλω να θυμίσω το εξής. Πρώτα, οι στόχοι της ανατολικής γειτονίας είναι ο πολιτικός διάλογος, η σύνδεση και οι οικονομικές σχέσεις πιο στενές. Δεύτερον, προφανώς μπορούν και βάσει του άρθρου 49 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να υποβάλουν αίτηση ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίω εφόσον ε, συμφωνούν με τις βασικές αρχές και αξίες. Τρίτον, αυτό απαιτεί ε, την τήρηση τη δημοκρατίας του κράτους δικαίου και των βασικών θεμελιωδών ελευθεριών. Αυτά είναι προαπαιτούμενα, τα οποία θα πρέπει να θυμίζουμε συνεχώς. Για την έκθεση, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία ήδη έχουν μια συμφωνία σύνδεσης και ε, μια διευρυμένη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξες και θέλουν να δουν και να μπορούν να κάνουν και άλλες πρόοδους. Αλλά κάθε πρόοδος θα πρέπει να αντανακλά και τις απόψεις κοινωνίας και όχι μόνο των κυβερνώντων. Και θέλω να τονίσω και να πω ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουν συμφωνία ε, σύνδεσης ή δεν επιθυμούν ε, κάνουν μεταρρυθμίσεις για μας. Αυτές οι χώρες δεν είναι εταίροι δεύτερης κατηγορίας, αλλά εξίσου σημαντικές, όπως και οι υπόλοιπε. Ε, στο εξή θα έχουμε τη συμφωνία με την Αρμενία, όπως ακούσαμε, και με το Αζερμπαϊτζάν ακόμα κάνουμε διαπραγματεύσεις. Η δική μου πολιτική ομάδα ε, έχει προσδοκίες από τη Σύνοδο Κορυφής του Νοεμβρίου. Αυτή η Σύνοδος θα καταγράψει την κατάσταση της τελευταίας διετίας και για τη δική μου πολιτική ομάδα έχει σημασία ε, τα αποτελέσματα που επιτύχαμε μέχρι τώρα ε, να είναι κατανοητά και ορατά προς την κοινή γνώμη, να τα γνωρίζει ο κόσμος και να τα μαθαίνει. Επίσης θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ποια είναι ε, τα καθηκόντα και υποχρεώσεις που μας περιμένουν. Δηλαδή υπάρχουν κάποια συμπεφωνημένα που δεν έχουν ακόμα ικανοποιητικώς εφαρμοστεί και υλοποιηθεί παντού. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα ούτε ικανοποιημένοι και οι δύο πλευρές με την υλοποίηση και την πρόοδο αυτής. Θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε τις συζητήσεις. Τι σημαίνει άραγε να πρέπει κανείς να προστατεύεται ε, και απέναντι στη Ρωσία και τι επιπτώσεις έχει αυτό για τη χώρα του καθενός. Πρώτο παράδειγμα. Μειονότητες. Σχολεία. Εκπαίδευση. Αν στην Ουκρανία το περιορίζουν μόνο στο δημοτικό στο μέλλον, τότε Μπορεί αυτό να μην αφορά τη Βουλγαρία, την Πολωνία και άλλες χώρες, αλλά μπορεί στο μέλλον να τις αφορά. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα και μόνο, ε, για να μην αναφέρω και άλλα. Αν δούμε τι γίνεται με τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Η δημοκρατία καμιά φορά είναι δύσκολο κεφάλαιο. Ακόμα και αν σε πρώτη γραμμή ε, σε, σε πρώτη φάση ε, έχουμε μια, μια συγκεκριμένη πελατεία. Τώρα εγώ δεν θέλω να χαρακτηριστώ foreign agent, έτσι ξένος πράκτορας, αλλά καταλαβαίνουμε για ποια πράγματα μιλάμε. Στη Μολδαβία, στην Ουκρανία και στη Γεωργία, αν μη τι άλλο. Τι νόημα λοιπόν έχει η ανατολική εταιρική σχέση ή τι στόχο έχει η ανατολική εταιρική σχέση. Διαφύλαξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας ε, με ε, τις ανατολικές μας ε, γειτονικές χώρες. Και μονίμως και όχι αναδιαιτία σε συνόδους κορυφής. Θα επιτύχει η ανατολική εταιρική σχέση μόνο εφόσον καταφέρουμε και εμείς και οι εταίροι να μεταφράζουμε στην πράξη τα όσα συμφωνούμε στις συνόδους κορυφής. Και τελειώνω λέγοντας ότι ορίσαμε ρητά θα πρέπει να υπάρχουν προοπτικές, όχι μόνο η απότερη προοπτική, αλλά και πιο κοντινές. Με συγκεκριμένα παραδείγματα, με θετικές κινήσεις, όπως είναι το Σέγγεν, ξέρω εγώ, και άλλες μορφές συνεργασίας. Αλλά η προϋπόθεση για να μην δημιουργούμε φρούδες ελπίδες είναι ότι όσα έχουμε συμφωνήσει μέχρι τώρα θα πρέπει να εφαρμόζονται για να έρθει και το επόμενο βήμα για το οποίο είμαστε νομίζω πρόθυμοι όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Κνούτ Φλέκενστάιν. Η κυρία Ανδρή Κέινε, Θέλετε να προσθέσετε τίποτα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κνούτ του Φλεκεστάιν για την εξαιρετική συνεργασία. Αυτή η προσπάθεια να έχουμε δύο συντάκτες από διαφορετικές πολιτικές ομάδες δεν είναι κάτι που ήθιστε εδώ και δεν είναι και απλό. Ωστόσο, ελπίζω ότι καταφέραμε να αφορούμε μια συμφωνία. Να ευχαριστήσω και τους κοιόδες εισηγητές για τη συνεργασία τους. 232 τροπολογίες κατατέθηκαν και σήμερα έχουμε 32 συμβιβαστικές ε, ε, τροπολογίες και μία προφορική που έχουμε συμφωνήσει ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πάνω από 90% από τις τοπολογίες που κατατέθηκαν καλύπτονται από τις συμβαστικέ. Δεν προβλέπω εκπλήξεις αύριο όταν θα ψηφίσουμε για αυτό το άγραφο. Αν και πρέπει ακόμα να δουλέψουμε με τον κύριο Φλέκεστάιν σε περίπτωση που κάποιες συμβιβαστικές δεν ψηφιστούν, δεν υπερψηφιστούν και θα χρειαστεί να ψηφίσουμε χωριστά στις ε, διάφορες τροπολογίες. Πρέπει εκεί να βρούμε συμφωνία για το πώς θα ψηφίσουμε. Ε, τώρα, όταν δει κανεί το σχέδιο και τις συμβαστικές, θα πρέπει να πω ότι μου αρέσει πολύ και τις εκεί συστάσεις και όχι πολλό μόνο επειδή είμαι συντάκτρια, μία από τις δύο συντάκτριες. Μου αρέσει επειδή αντικατοπτρίζει τις κύριες προτεραιότητες της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης. Μου αρέσει αυτό το έγραφο, λοιπόν γιατί είναι στραμμένο στο μέλλον, είναι ισορροπημένο και είναι και φιλόδοξο. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις τρεις χώρες εταίρους, Ουκρανία, Γεωργία και Μολδαβία. Και μια τέτοια πτυχή είναι η διαφοροποίηση που νομίζω επίσης είναι πολύ σημαντική. Η αρχή more for more και less for less θα πρέπει να εφαρμοστεί, θα πρέπει να γνωρίσουμε τις διαφορετικές ε, ε, διώξεις των εταίρων και η ανατολική εταιρική σχέση να είναι μεν για όλους, αλλά να έχει νόημα ε, και για τον καθέναν, γιατί δεν είναι όλα one size. Όταν είπα ότι είναι φιλόδοξο αυτό το σχέδιο, το είπα επειδή μιλάμε για το ε, ε, την, την εταιρική σχέση συν. Μιλάμε για χώρο Σέγγεν, μιλάμε για Ελληνική Ένωση, για Ενεργειακή Ένωση, για Ψηφιακή Ένωση. Όλα αυτά τα θέματα είναι τμήμα του, ε, τα, του εγγράφου μας. Οπότε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για τις τροπολογίες σας και ήταν πραγματικά μεγάλη μου ευχαρίστηση να δουλέψω για αυτό εδώ το σχέδιο. Ευχαριστώ και τους δύο και τώρα έχουμε σύντομες δηλώσεις των σκιωδών. Τσάλ Στάνοκ, θέλεις να πεις κάτι? Ναι, σύντομα πρόεδρε. Προφανώ είχαμε αυτή τη συζήτηση και παλιότερα και ήμουν παρόν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τι συμβιβαστικέ. Είναι κάτι με το οποίο είμαι πολύ εξοικειωμένο, γιατί και εγώ ήμουν εισηγητή πριν από μια δεκαετία για αυτή ακριβώ την έκθεση. Είναι κάτι που εν γέννη η ομάδα μου στηρίζει να αυξηθεί δηλαδή η δέσμευσή μα ε, όσο γίνεται περισσότερο επί τη βάση του μόρφο μόρ, όπω είπε και η κυρία Ανδριακένα. Το μόνο που μας απασχόλησε ήταν οι αρχές της ομάδας, των συμπροέδρων της ομάδας του Μίνσκ αναφέρεται στην δεφική αγκυριότητα και στο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση που είναι αντιπαρατηθέμενες αρχές στο διεθνές δίκαιο και η μία μπαίνει στα χωράφια της άλλης και αν θέλεις να βρεις λύση στο, στην ε, σύγκρουση Αρμενίας, Αζερβαϊτζάν και Ναγκόρνου καραμπα θα πρέπει να ληφθούν και τα δύο υπόψη. Αλλά να ε, υπερισχύσει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Εν γέννη είναι καλά δομημένη η έκθεση αυτή και σε μια χρονική στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ταλανίζεται από διάφορα σημαντικά θέματα όπως το Brexit, οι μεταναστευτικές ροές και οι κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν χώρες που έχουν μεγάλες ευρωατλαντικές ε, προσδοκίες, ε, ε, βλέψεις και αυτό είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αντιπροσωπεύει τη δημοκρατία, την ευμερία και την ειρήνη και ε, βεβαίως θα πρέπει να έχουμε ανοιχτό, να έχουμε προτάξουμε τη χείρα μας στις χώρες αυτές και στην ε, Αρμενία που πιέζεται από τη Ρωσία και που θεωρήθηκε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει με την DCFTA, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν θα μπορέσει να έχει μια πιο πολική, εξωτερική πολιτική που θα αναγνωρίζει το ρόλο και τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως η Ευρωασιατική Οικονομική Ένωση είναι σε ευρυκή κατάσταση για την ε, Αρμενία. Δεν Γιατί δεν χρειάζεται να έχει αυτή τη στιγμή από ένα πόδι σε κάθε πεδίο. Όπως η Γεωργία και η Ουκρανία και εμείς βεβαίως ε, έχουμε ιδιαίτερες επόψεις όσον αφορά την Ουκρανία και την ε, επεκτατική πολιτική της Ρωσίας εδώ, εκεί και εκεί θα επεκταθούμε όταν αυτό θα χρειαστεί. Ευχαριστώ, Χέλμουντ Σόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές ε, για την έκθεση αυτή που κατέθεσαν, διότι η κοινωνία πραγματικά παρακολουθεί αυτά ε, τα φαινομένα και τη Σύνοδο Κορυφής, όχι μόνο στις χώρες αυτές, αλλά και στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε ποιες είναι οι νέες θέσεις, τι κάνουμε ε, με τα ε, θέματα μεταξύ των κρατών ή στο εσωτερικό των κοινωνικών. Άρα, η αγρότησα, ο φοιτητής, ο ανθρακορίχος, θα αναρωτηθεί και τι νόημα έχει για μένα αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θέλω να αναφέρω δύο σημεία μόνο όπου εμείς έχουμε προβλήματα. Πιστεύω ότι η ανατολική γειτονία και η νέα πολιτική συν όσο σωστή και αν είναι και ανοίγει την προοπτική της ένταξης, αλλά νομίζω αποπροσανατολίζει ε, ε, από τις υποχρεώσεις που έχουμε από τα συμφωνηθέντα που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Θα πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι για να μας υποστηρίζει μαζικά και ο κόσμος και στα 28 κρατημέλη αλλά και στις κοινωνίες των ενδεχομένων ε, νέων υποψηφίων κρατών ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως είναι πολύ νωρίς αυτή η προοπτική. Θα δείξει. Επίση, θέλω να σε πιστήσω την προσοχή στο εξή. Ίσως πολιτική ομάδα έχουμε ως αρχή της πολιτικής μας και την αιρεσιμότητα, ιδιαίτερα στην μακροοικονομική βοήθεια για τις χώρες και της Ανατολικής Γειτονίας, διότι πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό που να είναι ορόσημο, που να μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει για πώς αλλάζουν οι πραγματικότητες και οι καταστάσεις. Και ένα δεύτερο που παραμένουμε επικριτικοί σε αυτό είναι απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν μπορούμε να υποδιόμαστε ή να υποκρινόμαστε. Ότι δεν έχουν προχωρήσει εξελίξεις. Χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό που θα δίνει και μια προοπτική για το πώς θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Τι θα γίνει, θα ανανεώνουμε συνεχώς τις κυρώσεις Υπάρχουν αρκετά άρθρα στη διεθνή οικονομική ε, βιβλιογραφία. Λοιπόν, θα πρέπει να καθίσουμε κάτω, να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, να βελτιωθεί η περίπλοκη σχέση που έχουμε με την Ρωσική Ομοσπονδία και που έχει και επιπτώσεις στην πολιτική γειτονία. Πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χέλμουντ Σόλτς. Δεν έχω άλλους ομιλητές. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό. Αύριο θα ψηφίσουμε σε 9 η ώρα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές που ήρθατε και καλή συνέχεια και καλή τύχη στο έργο σας. Στο καλό να πάτε. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, we then come to item... Συνάδελφοι, πάμε τώρα στο σημείο 6 και 7. Συμφωνεί με τη Νέα Ζηλανδία. Καταρχάς, 48 τροπολογίες. Τένοκ, Τάνοκ, συνομιλή ηγητής. Έχει καταθέσει και δύο συμβαστικές δύο προτάσεις συμβαστικών τροπολογιών. Του είναι το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ησυχία, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ, όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, κάντε το με ησυχία τάξη. Ναι, πρόεδρε. Και στην εργασία μεταξύ ΕΕ και των κρατών μελών της αφενός και της Νέας Ισλανδίας. Να πω ότι χαίρομαι τώρα που έχουμε αυτή τη συμφωνία με την Νέα Ισλανδία, άλλη μια χώρα της κοινοπολιτείας και έχει αλλάξει όνομα αυτή η συμφωνία, αλλά είναι παρόμοια στην δομή και στην αντίληψη με την SPA. Υπεγράφει λοιπόν αυτή η συμφωνία από την κυβέρνηση της Νέας και της εκπροσώπους Ένωσης πριν ένα περίπου χρόνο και είμαστε στην διαδικασία επικύρωση και πιστεύω ότι η πρόοδος αυτής της συγκεκριμένη συμφωνίας εξελίσσεται ομαλά χάρη επίσης και στην καθολική αποδοχή και υποστήριξη που θα τύχει η συμφωνία αυτή εδώ στο Κοινοβούλιο. Είχαμε 48 λοιπόν τροπολογίες και δύο συμβαστικές ρεκόρ χαμηλών μάλλον χαμηλό ρεκόρ και μας υπενθυμίζει αυτό το ότι η Νέα είναι από τους πιο εγγύς εταίρους μας όσον αφορά το κράτος δικαίου και πολιτιστικά επίσης μια χώρα που ορσιάζει πολλούς ε, δεσμούς με την Ευρώπη. Έχω καταθέσει πρόεδρε και δύο συμβαστικές, απλά και μόνο για διευκρινήσεις, επιφέροντας κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες και όχι τόσο για να βρούμε κάποια πολιτική συνεννόηση μεταξύ των μελών. Επίσης να πω ότι στην έκθεση χαίρομαι που υπάρχουν θετικές αναφορές στην Συμφωνία Ελεύθερων, Ελευθερών Συναλλαγών μεταξύ Ένωσης και Νέας Ζηλανδίας, δηλαδή η συμφωνία η οποία τρέχει παράλληλα με αυτή τη συμφωνία την οποία συζητάμε, η οποία είναι βέβαια κάτι το διαφορετικό για τη βελτίωση των εμπορικών δεσμών και νομίζω ότι θα πρέπει βεβαίως και αυτή να την υποστηρίξουμε παρόλο που κάποιοι ενδεχομένω να διαφωνούν. Χαίρομαι επίση που αναφέρουμε και το ρόλο της Νέας Ζηλανδίας, μια χώρα μικρή που παρόλα αυτά έχει ένα δυσανάλογα μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει για το μεγεθό της στα διεθνή πράγματα, στις διεθνεί υποθέσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με την Ένωση όσον αφορά τις επιχειρήσεις κατά των πειρατών, όπως κάποιες που κάναμε πριν από δύο χρόνια, όπως επίσης η καταπολέμηση της διεθνούς δημοκρατίας με στρατιωτική παρουσία στο Αφγανιστάν και να πω επίσης ότι υπάρχουν και διάφορες παραπομπές στο ρόλο των τωρινών της, Λανδ... Ε, της Νέας Ισλανδίας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για μια οικονομία με λιγότερες εκπομπές. Ρίξε λίγο άνθρακα. Από τότε που ξεκίνησα την συγγραφή αυτή της έκθεση στην Επιτροπή μας, είχαμε, έχουμε μεσολαβήσει και οι εκλογέ το Σεπτέμβρη στην Ισλανδία. Θα δούμε λοιπόν τώρα πώς θα σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση και ποια θα είναι γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα δεν έχουν απόλυτη πλειοψηφία. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια συμμαχία, ένας συνασπισμός με τους πράσινους της Ισλανδίας ή τον Ισλανδία first, τον Ισλανδία πρώτα. Αλλά αυτό είναι ευροσκεπτικιστικό κόμμα. Ήταν υπέρ του Brexit. Και είδα ότι είχαν λιγότερες ψήφους αυτή τη φορά. Βλέπουμε λοιπόν ο λακισμός να υποχωρεί σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν λοιπόν κάποιες, κάποια ιδιαίτερα προβλήματα στην έκθεσή μας. Έχουμε περισμένο αριθμό τροπολογιών και ελπίζω να έχω την υποστήριξη των συναδέλφων μας ήδη από σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Τσάλφ Στάνοκ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές Ουγγουριάνοφ, Ελκ και Κριστία από τους σοσιαλιστές Ουγγουριάνοφ. Σε λίγα λεπτά έτσι, ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ για τη θαυμάσια δουλειά. Είναι και φίλος και βεβαίως η έκθεσή του είναι καλή, συμμεριζόμαστε κοινέ αξίε με τη Νέα Ζηλανδία και ανήκουμε στην ίδια οικογένεια. Είναι λοιπόν απόλυτα φυσιολογικό με αυτέ τι ομοιότητε και αυτή τη φιλία να έχουμε μια ισχυρή οικονομική εταιρική σχέση. Η συμφωνία αυτή που θα ψηφίσουμε αύριο είναι απαραίτητο βήμα για την άναξη νέων εμπορικών διαπραγματεύσεων με τη Νέα Ζηλανδία για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Χαίρομαι που υπάρχει ισχυρή συνένεση μεταξύ των ομάδων του Κοινοβουλίου, ώστε η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ισλανδίας και Ένωσης να αποτελέσει ένα καλό σημείο κίνησης προς μια πλήρη Συμφωνία Ελευθερών Συναγωγών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ και του υπόλοιπου συναδέλφου και όδης για τη σαφή έκθεση και τις νομοδοτήσεις τους που καταθέσαμε πριν τις διακοπές. Αποβλέπουμε σε μια πιο φιλόδοξη συνεργασία και αυτό ήταν και το πνεύμα των τροπολογιών που καταθέσαμε. Είναι μονοούντες εταίροι η Ισλανδία και η Ένωση και η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης νομίζω θα επιφέρει στενότερη συνεργασία, βελτιώντα το διάλογο και βελτιώντα επίση και τη συνεργασία σε διάφορου τομεί. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι βέβαιο ότι με την ψήφο μα στην ΑΦΕΤ αύριο θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα και θα μεταβάσουμε ένα ισχυρό και ενδιαφέρον κείμενο στην Ολομέλεια και πάλι ευχαριστώ του συναδέλφου και όλους και τον συντάκτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και Χριστία. Δεν επιθυμεί το λόγο κάποιο άλλος από ό,τι βλέπω. Όχι. Αύριο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και κατά πάσα πιθανότητα στην Ολομέλεια συζήτηση και ψήφο τον Νοέμβρη. 8 και 9 σημεία τώρα. Πάμε καλά και από χρόνο. Καζακστάν, καταρχάς. Χαίρομαι που δεν υπάρχουν τροπολογίες κατά των συστάσεων της κυρίας Υπάρχουν 30 συμβαστικές και 148 τροπολογίες επίσης και πολλές από την Ίντερ. Κυρία Γιακονσάρη, έχετε το λόγο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο σου. 147 λοιπόν τροπολογίες, όπως είπα και εσείς πρόεδρε. Οι περισσότερες νομίζω περιλαμβάνουν τα θέματα που ενδιαφέρουν και απασχόλησαν τους συναδέλφους στην συζήτηση που είχαμε. Εκτός από θέματα εξωτερικής πολιτικής, πολλές τροπολογίες αφορούν συγκεκριμένες ανησυχίες για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιδών δικαιωμάτων στο Καζακστάν. Να τονίσω ότι το Κοινοβούλιο αναμένει από το Καζακστάν να επιδείξει βούληση για αυτά τα θέματα και να απελευθερώσει τους ακτιβιστές και συνδικαλιστές που αυτή τη στιγμή είναι φυλακισμένοι θα καταθέσω και μία προφορική τροπολογία στην συμβαστική 4, επειδή έχουν εξεχθεί τα πράγματα ευτυχώ. Ακούσαμε ότι τέσσερις από αυτούς τους ακτιβιστές ήδη απελευθερώθηκαν. Καλή είδηση αυτή. Να ευχαριστήσω και τους σκιωδείς μου, για την πολύ καλή συνεργασία. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος, αύριο θα ψηφίσουμε για το σύνολο αυτή τη έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αγία Κονσάρη. Ποιος επιθυμεί το λόγο προ το παρόν κύριο Κούκα από το, από το Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχά την συγγήτρια για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτή τη διαδικασία και του κοιόδης για τη θαυμάσια συνεργασία. Είχαμε πολύ καρποφόρες συναντήσει την περασμένη εβδομάδα των σκιωδών και χαίρομαι που οι θέσει τη ομάδα μου ληφθήκαν υπόψη. Τα πιο σημαντικά ζητήματα ήταν το να έχουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι εμεί συμφωνούμε με την συμφωνία αυτή, κάτι το οποίο αντανακλά και τι θετικέ εξελίξει που είχαμε στο Καζακστάν όσον αφορά την σχέση του με την Ένωση. Θεωρώ ότι αυτή η PCA πρέπει, αυτή η συμφωνία θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για βαθύτερε σχέσεις και εμπορικές και θεσμικές πολιτικές με το Καζακστάν, η Ένωση είναι ο πρώτος επενδυτικός και εμπορικός εταίρος του Καζακστάν και διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην διαφοροποίηση της καζανικής οικονομίας. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι αυτό θα βοηθήσει και το Καζακστάν να διαδραματίσει ένα πιο σημαντικό διεθνή ρόλο και να οδηγήσει σε ένα πυρηνικό αφοπλισμό. Γιατί έχουμε ακόμα μια χώρα η οποία είναι σημαντικό παίκτη στην Ασία και δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να θερύνουμε ο Καζακστάν συνεχίσει να δραματίζει σημαντικό επικοδομητικό ρόλο σε αυτό το πεδίο. Έχουμε εδώ λοιπόν το θέμα των ελευθεριών όπως ελευθερία έκφραση στα ΜΜΕ, συγκεντρώσεις λοιπά Έχουμε τις συστάσεις της Βενετίας, ε, έχουμε επίσης και την εφαρμογή των προεγραφών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο κράτος δικαίου. Σε γενικές γραμμές ενθαρρύνουμε πάντως παρά, τις, παρά τα κοινά και τις ελλείψεις ε, το Καζαστά να προχωρήσει και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε αρκετά ισορροπη Θα ήθελα λοιπόν να στήσω την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Κούκαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια και την πολύ καλή επικοδομητική της στάση σε αυτό το δύσκολο κατά τα άλλα θέμα. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνολική στρατηγική της έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ να έχουμε πιο στενές σχέσεις και εταιρικέ σχέσεις και συνεργασία με το Καζαχστάν. Η κατάσταση όμως παραμένει δυσμενής. Η οικονομική πρόοδος στο Καζαχστάν είναι πανταχού παρούσα, αλλά δεν συμβαδίζει με την πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το αντίθετο θα έλεγα. Θυμίζω ότι η ΜΚΟ Συμμαχία κατά των Βασανιστήριων κατήγγειλε 163 νέες περιπτώσεις βασανιστήριων από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2016. Περιορίζεται η ελευθερία της έκφρασης. 500 άτομα κρατούνται προσωρινά απλώς και μόνο επειδή ήθελαν να συμμετάσχουν σε μια ειρηνική διαδήλωση. Δύο ειρηνικοί ε, διαδηλωτές έχουν καταδικαστεί σε πενταετή φυλάκιση απλώς γιατί βγήκαν στο facebook και σε κάποιες άλλες πλατφόρμες και εξέφρασαν την κριτική τους. Συνοψίζω. Καλό είναι και πολύ σημαντικό να έχουμε σχέσεις ε, και ε, βορείο με το Καζαχστάν ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρειάζεται προσοχή. Δεν θα πρέπει να ανοίξουμε όλα τα χαρτιά μας, να βοηθήσουμε και να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπόχνα για την ομιλία σας. Δύο ακόμα συναδέλφους έχουμε. Θα κλείσω όμως τον κατάλογο. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ και η δική μου πολιτική ομάδα θα στηρίξει την έκθεση αυτή. Είναι καταπληκτική έκθεση. Πάνω από 10 χρόνια ε, πριν ήμουν εγώ εισηγητής, δείχνει και πόσο καιρό είμαι εδώ βουλευτής. Και τότε η ανατολική γειτονία ε, δεν συμπεριλαμβάνει το Καζακστάν και εγώ το πρότεινα. Ε, έχουν ένα μικρό κομμάτι γης που γεωγραφικά ανήκει στην Ευρώπη πάνω από την Κασπία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η χώρα, τεράστια, έχει τεράστια κοιτάσματα ε, φυσικών ε, πόρων, αλλά είναι και ένα μοντέλο επιτυχές ε, ειρηνικής ευημερούσας κοινωνίας, όπου συμβιώνουν μουσουλμάνοι, χριστιανοί και πολλές άλλες μειονότητες γλωσσικές, εθνικές και θρησκευτικές. Με αγαστό τρόπο, καταπληκτικό συμβιώνουν. Αυτό είναι ενδεχομένω μια σοβιετική κληρονομιά και μπορεί να είναι και ένα παράδειγμα για τη Δύση, για το πώ μπορεί κανείς να συμβιώσει με άλλους πολιτισμούς, θρησκευτικέ κοινότητες σε μία χώρα. Εμείς θα πρέπει να τίνουμε χείρα βοηθείας προς το Καζακστάν, να δούμε τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια, να μελετήσουμε την κατάσταση, για πώς έχουν εξασφαλίσει μια τόσο αρμονική συμβίωση με πάρα πολύ μικρή ε, ριζοσπαστικοποίηση του Ουσμπεκιστάν έχει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από το Καζακστάν. Βεβαίω παραμένει πρόβλημα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακούσαμε, αλλά και τα εργατικά, εργασιακά δικαιώματα. Είναι και πολύ ψηλή η διαφθορά. Με αυτή την επιφύλαξη όμως μπορούμε να πούμε ότι το Καζακστάν είναι μια χώρα θαυμάσια, εκπληκτική και καλό θα ήταν να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό. Και εδώ και πολλά χρόνια το έχω πει και έχει πολύ ε, ε, ελπιδοφόρο και υποσχόμενο μέλλον. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Ρωσία έχει σημασία αυτό. Προσπαθήσει λίγο να ε, εναρμονίσει ε, τη, τους δασμούς του με τον ΠΟΕ ανεξαρτήτως συμφωνίας που έχει κάνει με την Ευρωσια... Ε, Ευρωσιατική Ένωση. Και μπορεί να είναι και ένα είδος ε, ενδιάμεσης χώρας ανάμεσα σε εμάς και στη Ρωσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σπέιτ. Και η ομάδα ALDE υποστηρίζει αυτή την ενέκθεση. Νομίζω πως υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με, τον, ε, με το Καζακστάν και από την άλλη πλευρά με την στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί όπου βλέπουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Αλλά συμφωνώ ότι σε σχέση με άλλες χώρες της περιοχής, οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και το Καζακστάν αναπτύσσονται καλά, γιατί και οι δύο πλευρές ενδιαφέρονται γι' αυτό. Και επίσης ε, η ανάπτυξη του Καζακστάν, ειδικά στον οικονομικό τομέα, είναι εξωσημείωτη. Ταυτόχρονα θα ήθελα να τονίσω τη σημασία για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Καζακστάν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε κάποια ονόματα σε αυτό το σχέδιο έκθεσης, αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλοι για τους οποίους ανησυχούμε, ας πούμε, συνδικαλιστές, ο κύριος Νόρφεκ και ο κύριος Βάγεφ που έχουν καταδικαστεί. Βλέπουμε λοιπόν ονόματα στο σχέδιο εκθεσή μα που δεν καλύπτουν 100% όλων μας των ανησυχιών και προβλημάτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά συνοψίζοντα ελπίζω πως το Καζακστάν θα δει την έκθεσή μας και την ε, ε, διάθεση της Ένωσης να προχωρήσει στη σχέση μας. Θα δει εκεί λοιπόν ένα μήνυμα καλής θέληση. Επίσης, τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, θα τα τονίσουμε ώστε το Καζακστάν να ελπίζουμε να ανταποκριθεί με θετικό τρόπο και γρήγορα. Ευχαριστώ, κύριε Πάιτ. Άλλα σχόλια. Όχι, ούτε η συγκεκριτή θέλει να κλείσει. Η συγκεκριτή, συγγνώμη. Ωραία λοιπόν, αύριο θα εξετάσουμε ξανά το θέμα και η ψηφοφορία θα γίνει μάλλον τον Νοέμβριο. Σας ευχαριστώ. Πάμε στο σημείο 10. Βίγκαν. Είναι στο δρόμο. Άμα δεν είναι εδώ ο κύριος Βίγκαν δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε. Οπότε θα περιμένουμε λίγα λεπτά. Αναγκαστικά. Καλύτερα να μείνετε εντός αιθούσης. Παρακαλώ να σημειώσετε το σημείο 10, είναι και κλεισμένο των θυρών συζήτηση. Όλοι όσοι δεν ε, πρέπει να μείνετε ε, μπορείτε να φύγετε από τώρα.